παρούσες ε, συνεδρίασεις θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περίοδου συνόδου. Αν δεν υπάρχουν ε, σχόλια, επί των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν σήμερα θα απευθυνθούν εκεί όπου προορίζονται. Έτσι ολοκληρώθηκαν ε, οι σημερινές μας εργασίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Καλό ταξίδι.